Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Εντάξει, πέμπτη είναι, το ξέρω. Όλοι θέλουν να προλάβουν αεροπλάνα και τρένα. Πάμε λοιπόν. Να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες μας. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση αρχικά. η οποία έχει ως εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 166 του κανονισμού, ο πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει ποινή στον κύριο Ντεκράφ για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της 28 Οκτωβρίου 2015. Ε, ε, αυτό αφορά πενθήμερη αποζημίωση ε, και ε, είναι γνώση ε, του κυρίου Τεγράφη απόφαση αυτή για πενθήμερη ε, παρακράτηση αποζημίωσης. Now, I will... Λοιπόν, θα μιλήσω ρωμανικά. Τώρα έχω λάβει από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών